κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 16, αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 18, αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 29, το αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. Παράγραφο 30, αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, απόχέ. εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, Αποχέ εγκρίνεται. 34, αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, απόχέ. εγκρίνεται. Το πρώτο τμήμα, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά,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 Απορρίπτεται. Παραγραφός 38, αρχικό κείμενο, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 7, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 56, το αρχικό κείμενο, σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, υπέρ, έναξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι.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 29 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική αναφορά 43 υπέρ κατά αφορές εγκρίνεται. Αιτιολογική αναφορά 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη ψηφοφορίας.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 Παράγραφος 44, ονομαστική ψηφοφορία του αρχικού κειμένου. Μάλλον επαληθεύουμε την τροπολογία 10. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την τροπολογία 10 έναρξης ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 44, ονομαστική ψηφοφορία έναρξης ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 46 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 56. Το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 70, αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη ή ε, τροπολογία 1 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 5 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Στο, φτάνουμε στο ψήφισμα ε, της Επιτροπής ΑΦΕΤ στο σύνολό του, ε, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση Donjon. Τροπολογία 18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 3 αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 21, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 23, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι, λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο της παραγράφου 12 σε τρία τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη τη ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 σε δύο τμήματα και τα δύο σε ονομαστικές ψηφοφορίες. Πρώτο τμήμα, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Ε, λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο της παραγράφου 16 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Ε, ονομαστική ψηφοφορία, μάλλον έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο της παραγράφου 21 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αποχές επαλήθευση έναξης ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 31 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 ονομαστική ψηφοφορία έναξης ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο της παραγράφου 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 26. Αρχικό κείμενο. Ονομαστική ψηφοφορία. Άνοιξη ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Ονομαστική ψηφοφορία. Έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 37. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία. Ένάξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφο 43, το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 48, τροπολογία 32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφο 48, αρχικό κείμενο, ονομαστική ψηφοφορία, έναξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. τροπολογία 39 υπέρ. Κατά. Παρακαλώ άλλη μια φορά. Τροπολογία 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Ονομαστική ψηφοφορία. Έναξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Παράγραφος 64. Αρχικό κείμενο. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 66, αρχικό κείμενο, ονομαστική ψηφοφορία, έναξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 68, αρχικό κείμενο, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 69, αρχικό κείμενο, ε, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Παράγραφος 69. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Παράγραφος 73. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 38. Ονομαστική ψηφοφορία. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο. Καταπίπτει. Τροπολογία 15. Ονομαστική ψηφοφορία. Αναξή της ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 35, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 17, υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. Παράγραφος 106, αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 107, αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 111, αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη τη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Το ψήφισμα στο σύνολό του όπως τροποποιήθηκε ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε για να ολοκληρώσουμε στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Ονομαστική κλίση για την τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρασε. Απορρίπτεται. 17 ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 36 ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 37 Ονομαστική κλίση, άρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 1. Ονομαστική κλίση, άρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρας απορρίπτεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19 ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41 ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. έγκριναν. 42 υπέρ. Κατά. απόχέ Απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. απόχέ, Απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο για την παράγραφο 7 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο στην παραγραφό 8, ονομαστική κλίση, άρχιτη ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Εγκρίνεται. 3. Τροπολογία 3. Ονομαστική κλίση, άρχιτη ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Απορρίπτεται. 46. Ονομαστική κλίση, άρχιτη ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρας. Απορρίπτεται. Πέραγραφος 9 αρχικό κειμένο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δύο, δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, παράγραφος 10, ονομαστική κλίση, έρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Απο... Ε, πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 48. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. 71. Ονομαστική κλίση έρχεται ψηφοφορία. Έψηφισαν απαντέ. Πέρας. Εγκρίνεται. 49 ονομαστική κλίση έρχεται η ψηφοφορία. Έψηφισαν ε, άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 75 ονομαστική κλίση έρχεται η ψηφοφορία. Έψηφισαν ε, άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέσσερα τροπολογία τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 72 ονομαστική κλίση. Να ελέγξουμε για την 69. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. πέρα, Εγκρίνεται. 72 να μας εκκλησία έρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. πέρα. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο, ε, το έχουμε ολοκληρώσει 52 να μας εκκλησία έρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες πέρας. Απορρίπτεται. 74 ονομαστική εκκλησία έρχεται η ψηφοφορία. Έψηφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 70 ονομαστική εκκλησία έρχεται η ψηφοφορία. Έψηφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται αρχικό κείμενο, ε, το έχουμε ολοκληρώσει. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 73 ονομαστική κλίση έρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 54 ονομαστική κλίση έρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας απολύτω. 76. Νομίζω είχε κάποιο σου πει ότι έχει προφορική τροπολογία. Κύριε Φρόιτ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ήθελα μια προφορική τροπολογία να υποβαλώ. Το Στρασβούργο θα κατασταθεί από Βεξελίσσα. Δηλαδή, ε, η πλειονότητα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων να λέει η φράση. Είναι σημαντικό για του Ευρωπαίου πολίτε να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι απόψει του και οι αγορέ, δηλαδή το τόπο συζήτηση των Ευρωπαίων πολιτών να, γίνεται στις Βρυξέλλες, να οργανωθεί στι Βρυξέλλε και όχι στο Στρασβούργο. Ε, συνάδελφε Φρόιντ, δεν χρειάζονταν όλη αυτή η αιτιολόγηση. Υπάρχουν αντιρρήσει για αυτήν την τροπολογία. 40 συνάδελφοι τουλάχιστον. Έχουμε 40, οπότε δεν μπορούμε να δεχτούμε την προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε την αρχική εκδοχή του, ε, της τροπολογίας 76. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18 αρχικό κειμένο σε με τα πρώτα τμήμα ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 57 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 60, ονομαστική κλίση, έρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν πάντες πέρας. Απορρίπτεται. 61, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 62, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 63, ονομαστική κλίση, έρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες πέρας. Απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 ονομαστική κλίση έρχεται ψηφορία, Εψήφισαν άπαντες πέρας. Απορρίπτεται. 65 ονομαστική εκκλησία έρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5. Ονομαστική κλίση έρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 26. Ονομαστική κλίση έρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67. Ονομαστική κλίση έρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29 ονομαστική κλίση έρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7 υπέρ. Ονομαστική κλίση, συγγνώμη, άρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν Απάντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9. Ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. πέρα, Απορρίπτεται. 10. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. 33. Ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. πέρα. Απορρίπτεται. 11. Ονομαστική κλίση άρχιτη ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Απορρίπτεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 13. Ονομαστική κλίση άρχιτη ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Απορρίπτεται. 14. Υπέρ. Κατά. Από 15 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 34. Ονομαστική κλίση έρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. πέρα. Απορρίπτεται. 35. Ονομαστική κλίση έρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. πέρα. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το ψήφισμα όπως τροποποιήθηκε συνολικώς, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες πέρας. Εγκρίνεται. Ich danke Ihnen sehr. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, να φύγετε από την αίθουσα ήσυχα. Θα ξεκινήσουμε τις επεξηγήσεις ψήφου. Θα περάσουμε λοιπόν σε επεξηγήσεις ψήφου. Λέει πρόεδρος σε πολλές γλώσσες. Please, colleagues, leave the room in a quiet manner. Αποχωρείτε ησύχως. Τάικοστατομ önöket, hogy a sok szóbeli szavazat indoklási kérelmet Λόγω του μεγάλου αριθμού των επεξηγήσεων ψήφων και επειδή είχαμε και πολλές ψηφοφορίες θα πρέπει να ολοκληρώσουμε στις 14 και 45. Οπότε θα πρέπει να είστε έτοιμοι ε, για να τηρήσετε το χρόνο ομιλία. ό,τι δεν προλάβουμε σήμερα θα ολοκληρωθεί αύριο. Ή μπορούν να αποσταλούν και γραπτός όσοι δεν προλάβουν να πάρουν το λόγο. Συνάδελφοι, ξεκινούμε τις επεξηγήσεις ψήφου. Ψηφίζουμε για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ο κύριος Κέλαχαν. Κέλεχα από του Ρινιού. Με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία όλα τα κράτη-μέλη θα μπορούν να περνούν σε μια κοινωνία με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό όμως είναι απλώς η αφετηρία. Παρακαλώ, θα περιμένουμε 30 δευτερόλεπτα για να αποχωρήσουν όλοι και μετά θα ξαναρχίσετε. Θα σας ξαναδώσω το λόγο, διακόπτη πρόεδρος. Δεν ακούω καν τι λέω, λέει ο μιλητή. Και τώρα έχετε το λόγο. Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα επιτρέψει σε όλα τα κράτη-μέλη να περάσουν σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών. Αυτό είναι απλώς η αφετηρία όμως. Ψήφισα υπέρ τη συμφωνίας αυτής, γιατί είναι ένα καλό σχέδιο για να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να κάνουμε τα εξής πράγματα. Πρώτον, θα πρέπει να υποστηρίζουμε τις κοινότητες για να υπάρχει μια δίκαιη μετάβαση προς τις χαμηλές εκπομπές. Δεύτερον, θα πρέπει οι κυβερνήσεις να είναι διατεθειμένες να πάρουν σκληρές αποφάσεις τώρα, όχι αργότερα. Και τρίτον, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι επιχειρήσεις συνεργάζονται με τις κυβερνήσεις, γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο για να σώσουμε τον πλανήτη. Οι φρικτές πυρκαγιές στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή θα πρέπει να μας φοβήσουν όλους εδώ στην αίθουσα. Στη χώρα μου έχουμε επίσης ε, ακραία καιρικά φαινόμενα. Επίσης θα πρέπει να δώσουμε ελπίδα στους λαούς ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί χωρίς την ελπίδα οι άνθρωποι θα παραιτηθούν. Θα ήθελα να παρακολουθήσετε όλη την ομιλία του Νεοζηλανδού Πρωθυπουργού, της Νεοζηλανδού Πρωθυπουργού πριν τα Χριστούγεννα, που με γέμισε ελπίδα. Ελπίζω, αν τα κάνουμε όλα αυτά, να σώσουμε τον πλανήτη. Συνάδελφε, προσπαθήστε απλώς να τηρείτε το χρόνο του ενός λεπτού. Διότι θα πρέπει να κόβω το μικρόφωνο. 60 δευτερόλεπτα. Έχουμε 60 λεπτά για όλο, για όλο το γύρο των επεξήσεων. Είναι η πιο σημαντική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα λάβει ποτέ στην ιστορία της. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία σηματοδοτεί τις απαραίτητες προσπάθειες που πρέπει να γίνουν για να προστατεύσουμε το πλανήτη και να προστατεύσουμε την βιοπικιλότητα. Ένα πλαίσιο δράση θα πρέπει να συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η ρήπανση ποτέ δεν σταματά στα εθνικά σύνορα. Αφορά κάθε πολίτη και κάθε κοινότητα και πρέπει να δράσουν όλοι και στην περιοχή μου έχουμε τριπλάσια ρήπανση από το ανώτατο επιτρεπτό όριο. Παρ' όλα αυτά, ο Πρωθυπουργό μα επιτρέπει τη ρήπανση να κάνει τη δουλειά τη. Οι τοπικέ ε, κοινότητε προωθούν τα δικά του προγράμματα. Παραδείγματο χάρη, εμεί γίναμε μια πόλη χωρί πλαστικά. Η νέα συμφωνία ξέρει ότι η κατάσταση αυτή βλάπτει τον πλανήτη και υποσκάπτει το μέλλον των μελλοντικών γενεών. Θα πρέπει να δράσουμε τώρα. Πρόεδρος. Η κυρία Τζόνς, ένα λεπτό παρακαλώ. Mrs. Jones, the floor is... Έχετε το λόγο. Κυρία Τζόνς. Ευχαριστώ. Η κλιματική αλλαγή και τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι η μεγαλύτερη απειλή της ανθρωπότητας και θα πρέπει να πολεμήσουμε. Η Ευρώπη χρειάζεται ένα νέο βιώσιμο οικονομικό μοντέλο κατάλληλο για την δεκαετία 2020. Θα πρέπει τα, η κοινωνική και η περιβαλλοντική πρόοδος να συνδυάζονται. Γιατί οι ανισότητες ε, είναι κατά της ευμερίας όλων και αφορούν όλους μας. ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αφορά όλη την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη Ρουμανία προς την Ιρλανδία. Το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι μια μεγάλη μάζα γης, θα πρέπει να δράσει και αυτό, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή. Εμείς ήμασταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που δηλώσαμε ότι υπάρχει κρίση κλιματική και θέλουμε να συνεργαστούμε τους ε, γείτονές μας και πρέπει να το κάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να αφορά όλη την Ευρώπη για την ευημερία και το καλό όλων. Είμαστε ηγέτε ε, στην κλιματική αλλαγή και η Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι περιβαλλοντικέ και κοινωνικέ πολιτικέ αναπτύσσονται για να εξασφαλίσουν τη δίκαιη μετάβαση και να υπάρξει δίκαιη οικονομική και κοινωνική και περιβαλλοντική αλλαγή. Θα πρέπει να, το, να κάνουμε ό,τι πρέπει, αυτό που απόκειται στο καθένα, είτε είμαστε εντό είτε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Μανουέλ Μπομπάρ. Συνάδελφοι, πρόεδροι, το Κοινοβούλιο δήλωσε πριν από λίγο την κατάσταση έκτακτης ανάγκης των το περιβάλλον και την οικολογία. Είναι απαραίτητο να δράσουμε τώρα, μια και είναι τόσο κατεπήγον αυτό το θέμα και προκηρύξαμε, το προκηρύξαμε και το δηλώσαμε όλοι μαζί. Το κείμενο που ψηφίσαμε έχει ενδιαφέρουσες προθέσεις, αλλά δεν παίρνει τα απαραίτητα μέτρα με βάση το, τα προβλήματα. Ο στόχος μείωσης 50% των ε, εκπομπών του αερίου θερμοκηπίου ήταν κάτι που το είχαμε αποφασίσει και στην προηγούμενη νομοθετική ε, θητεία. Θα πρέπει να φτάσουμε στο 65% μέχρι το 2030, αν θέλουμε να μειώσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας. Χρειάζονται απαραίτητε μεταρρυθμίσεις τη κοινή γεωργική πολιτική. Ενώ το κείμενο που παρουσίασε η Κομισιόν δεν μας επιτρέπει να περάσουμε στην οικολογική μετάβαση της γεωργίας. Το κείμενο δεν καταγγέλει τις εμπορικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Για όλα αυτά τα σημεία το κείμενο είναι επαρκές. Επομένως δεν μπορώ δυστυχώς να το υποστηρίξω. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Στίγκριτ. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Αρχίζει αυτή η διαδρομή, αλλά είναι κάτι σαν η Ευρώπη να πηγαίνει να Μεγάλα λόγια από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν χωρίς να μας λέει όμως πώς θα γίνουν όλα αυτά, ποιες θα είναι οι συνέπειες και ποιος θα είναι ο αντίκτυπος. Ε, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, λαϊκισμός είναι. Διότι επενδύσεις σε έναν τομέα σημαίνει έλλειψη επενδύσεων σε άλλον τομέα. Χιλιάδες ε, δισεκατομμύρια σε μέτρα για το κλίμα χωρίς επενδύσεις ε, στην ε, νοσηλεία ή άλλους τομείς ε, δεν ε, θα αποτελέσουν καλή βάση για το μέλλον. Και βλέπουμε έτσι ότι η φιλοδοξίες σας ε, για το φεγγάρι ε, ε, δεν σημαίνουν τίποτα. Θα πρέπει να έχουμε ρεαλιστικούς στόχους και να είναι σαφείς οι συνέπειες. Γι' αυτό καταψηφίζω την πρόταση του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ, Σόιτροβα, από το ΕΛΚ. Κυρίες και κύριοι, η τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη νέα πράσινη συμφωνία είναι πολύ σημαντική, φιλόδοξη, περίμενα, λογική. Βέβαια δεν είναι τόσο λογική, περισσότερο φιλόδοξη όταν έγινε η ψηφορία εγώ απέσχον και εστίασα την προσοχή μου σε δύο σημεία. Πρώτα-πρώτα στη Γεωργία, διότι χρειαζόμαστε βιωσιμότητα και στη Γεωργία και επίσης θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι αυτό μπορεί να το πετύχουμε όταν δώσουμε κίνητρα εις τους αγρότας. Και θα μπορούσαμε να πληρώσουμε τις προϋποθέσεις και τους όρους της νέας συμφωνίας. Να δώσουμε επόμενος νέες ευκαιρίες ούτως ώστε να καταβολήσουμε την κλιματική αλλαγή, Γεωργή. Οπότε σε αυτό το μέτωπο η πρόταση είναι θετική, αλλά δεν αποδέχομαι μία τροπολογία. Εκεί που μιλάει για την πυρηνική ενέργεια. Επίσης, αναγνωρίζεται η επικουρικότητα και τότε τα κρατημέλη μπορούν να χαράξουν το δικό τους ενεργειακό, ενεργειακή πολιτική, ενεργειακό μείγμα. Οπότε αυτή η τροπολογία, την πυρηνική ενέργεια είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό και απέσχον. Η κυρία Γιώβεβα έχει το λόγο. Εγώ υπερψήφισα το ψήφισμα για την Πράσινη Συμφωνία διότι αντικατοπτρίζει ε, τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλουμε ε, ουδετερότητα όσον αφορά τον άνθρακα, θέλουμε ε, υψηλό βιωτικό επίπεδο ε, σε όλον τον πλανήτη. Πρόκειται για ισορροπημένη πρόταση και θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα της αλλαγής του κλίματος και να έχουμε δίκαιη μετάβαση και να δημιουργήσουμε νέε δυνατότητες. Πολύ σημαντική είναι η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών ε, και τον οικονομικό τομέα. Θέλουμε λοιπόν ε, μία ουδέτερη ως προς άνθρακα κοινωνία και θέλουμε να καλέσουμε και το υπόλοιπο του κόσμου να συνεργαστεί. Είναι απαραίτητη η Πράσινη Συμφωνία ε, ταυτόχρονα αποτελεί ευκαιρία. Θα μπορέσουμε έτσι να συνεργαστούμε και με άλλους παράγοντες για να εμποδίσουμε την αλλαγή του, του κλίματος. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, λέει ο κύριος Πόλτσακ. Εγώ τοποθετήθηκα υπέρ, διότι είναι η σωστή κατεύθυνση που πρέπει να την πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είναι η πρόκληση πολύ σημαντική αλλά είναι και για την Τσεχία μια που έχουμε ακόμα κάποιες περιοχές, περιφερειές της χώρας δεν είναι έτοιμες για αυτήν την αλλαγή και να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε τάξει είναι μια πρόκληση για να εξυγχρονίσουμε την οικονομία αλλά, αλλά εγώ θεωρώ ότι το πράσινο φως που δόθηκε σε κάποια σημεία και κάποιες τροπολόγες δεν είναι τόσο χρήσιμες γιατί είναι περίεργο να μην θέλει να υπάρχει απαρίθμηση στο Κοινοβουλίο όσον αφορά τα σχετικά μέτρα των επιπτώσεων ε, για εμένα αυτό ήταν απογοητευτικό και κανονικά θα είχα απόσχει αλλά δεν ήθελα να τοποθετηθώ αρνητικά και τελικά ψήφισα υπέρ οπότε θα πρέπει να μην ξεχνούμε πόσο βλάπτουμε τον πλανήτη και θα πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Πρόεδρος. Charlie az ECR-tól. Ευχαριστώ. Βέιμερς από το ECR. Όχι, Βερόνικα Βρετσιόνοβα. Ζητώ συγγνώμη, λέει η πρόεδρος. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο, λέει η κυρία Βρετσιόνοβα. Εγώ δεν ψήφισα υπέρ αυτού του κειμένου. Πάντως, συμφωνώ με κάποιους στόχους όπως τον να προαγάγουμε την βιοπικιλότητα, να αυτοδεύσουμε τα δάση κλπ. Πάντως υπάρχουν κάποια σημεία που είναι πάρα πολύ ακραία που δεν θα είναι δόκιμα, δεν θα πετύχουν το στόχο και θα είναι αντίθετα πάρα πολύ επαχθή για τον κόσμο. Και Ρώτησα τους ψηφοφόρους μου αν συμφωνούν με το υψημένο κόστος ενέργειας και θέρμανσης. Εσείς ρωτήσατε, ρωτήσατε αν δέχονται ψηφοφόροι το πλήγμα στην απασχόληση. Μην κρύβετε από τον κόσμο το τι αποφασίζεται σε πολλές χώρες έχουμε τέτοια αρνητικά φαινόμενα και έχουν ανέβει οι τιμέ. Ο πλευρά των Πρασίνων. Τώρα, Φίλιπ, ένα λεπτό. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση τώρα. Η νέα πράσινη συμφωνία είναι πάρα πολύ σημαντική πολιτική, έτσι θα μπορέσουμε κάτι να κάνουμε, να έχουμε λιγότερη ανισότητα και να γίνει αυτό ο μετασχηματισμό με το μηδενικό άνθρακα στην Ευρώπη και γι' αυτό και είμαι περήφανη. Ήταν πολύ σημαντική ψήφο που ρίξαμε εμεί οι πράσινοι. Το κοινοβουλίο επιτέλου κάτι κάνει και έτσι σιγά σιγά να σταματήσουν τα ρηχτά καύσιμα και θα εξασφαλιστεί ότι και οι γυναίκε θα καλύπτονται από τη νέα συμφωνία. Όμως η διαδρομή αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί. Εμείς οι πράσινοι θα συνεχίσουμε, θα πιέζουμε την Επιτροπή να υλοποιήσει πραγματικά την Πράσινη Συμφωνία και από κοινωνική πλευρά και από περιβαλλοντική. Πάρα πολύ σημαντικό είναι να στατευτεί και ο κόσμο για αυτή την προσπάθεια μέσω φορέων κοινωνικών. Γόλα. Και εσεί, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε διάφορα θετικά σε αυτό το κείμενο. Ας πούμε, το 20 λέει για το κόστος της καινοτομίας που δεν πρέπει να το φέρνουν οι πιο φτωχοί, την κυκλική οικονομία, τα μικροπλαστικά. Πολύ πολύ καλά να αυτά και για την αναβάθμιση των εργασιακών ε, διατάξεων, αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω συνολικά γιατί υποβαθμίζεται ε, ο καρδιά του κατεπήγοντος και ε, συνεχίζονται οι ανοσότητες, το Μερκοσούρ, τίποτα, ε, λέει και για το φυσικό αέριο τρελά πράγματα που το προωθεί και τα όσα λέει για την Γεωργία. Εγώ νομίζω ότι η κοινή η πολιτική βλάπτει και πολύ. 60 δις δαπανώνται από τις τσέπες των φορολογουμένων επιδοτήσεις κλπ. Και όλα αυτά είναι για μεγάλο ε, επιχειρήσεις ε, και όχι υπέρ των μικροκαλλιεργητών. 55% λέει το κοινοβούλιο, μέχρι το 2030 πρέπει να έχουμε κατέβει σε εκπομπές και θα πρέπει όλα αυτά να περάσουν και από μελέτη επιπτώσεων. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κλέρ Ντέιλι είναι η επομένη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε ενώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα πάμε καλύτερα από άλλε οικονομίε του κόσμου όσον αφορά την αντιμετώπιση του θέματο του κλίματο, δεν σημαίνει ότι είμαστε αρκετά καλοί. Ε, καταψήφισα το ψήφισμα, διότι ε, δεν είναι επαρκέ ε, όσον αφορά τα όσα πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Κάποιες ε, από τις ψηφοφορίες των τροπολογιών μας έδειξαν ε, ότι πολύ μιλάμε, αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Η απόρριψη της τροπολογίας που κατονομάζει τις 100 ε, μεγαλύτερες εταιρείες που είναι υπεύθυνε για το 75% των εκπομπών, το ότι μιλάμε για δίκαιη μετάβαση, αλλά χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερα χρήματα για να επιδοτούμε δραστηριότητες ε, ρηπογόνε το ότι ε, δαπανούμε δισεκατομμύρια ε, στην βιομηχανία άμυνας που αυξάνει κατά πολύ το οικολογικό μας αποτύπωμα. Όλα αυτά δείχνουν πόσο επίγοντα είναι αυτά που πρέπει να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Γκλουικ από το Renew. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω γερμανικά. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι. Δεν συμφωνούμε με όλα που συμφωνήθηκαν και αποφασίστηκαν σήμερα για την απόφαση για την Πράσινη Συμφωνία. Παρ' όλα αυτά δεν θα την απορρίψουμε. Δεν θα το απορρίψουμε το ψήφισμα, διότι ως άμεσα αιρετή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είμαστε αυτοί που πρέπει να υπερασπίσουμε το κλίμα και το περιβάλλον. Αυτό το πιστοποιητικό το ευρωπαϊκό που αφορά την κίνηση και τα οχήματα και τα κτίρια δεν το καταλαβαίνουμε. Όλοι οι τομείς που, ε, τους οποίους αφορά το πιστοποιητικό αυτό θα επιτύχουν τους στόχους όσοι δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το πιστοποιητικό δεν θα τους επιτύχουν. Έχουμε ένα πολύτιμο εργαλείο κατά την άποψή μας με αυτό το πιστοποιητικό ακόμη και στους τομείς ε, της θέρμασης κτηρίων όσο και, της, ε, ε, και των οχημάτων. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής ο κ. Γιώργης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα ψηφίσουμε υπέρ της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας γιατί θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη. Είναι απαραίτητη η Πράσινη Συμφωνία χωρίς ε, αλληλεγγύη και χωρίς την κοινωνική διάσταση. Θα, ε, δεν θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τους ανθρώπους. Ε, αν η πράσινη αυτή συμφωνία ωφελεί μόνο λίγους ενώ το κόστος το μοιράζονται όλοι, τότε είναι σαφές ότι θα υπάρξουν διαμαρτυρίες. Έχουμε όμως ακόμη χρόνο για να διορθώσουμε την κατάσταση και μάλιστα με ψήφισμα σχετικά με την κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Ε, Ευχαριστούμε επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό. Ε, Μέλλερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε εδώ πόσο αποφασισμένοι είμαστε ούτω ώστε να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή τη μάχη υπέρ του περιβάλλοντο. Αυτό είναι αναπόφευκτο και σημαντικό για τον άνθρωπο και για τη βιοπικιλότητα. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι κάθε οικολογικό θέμα είναι τόσο δεσμευτικό για τι εθνικέ κυριαρχέ πολιτικέ και το ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε τι εξουσίε που παρέχει αυτό το κείμενο, απολυταρχικέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υπερασπίζουμε ιδεολογίες γραφειοκρατίας ε, ε, σε ολόκληρο το κείμενο ουσιαστικά με διάφορα υπονοούμενα. Εμεί προτείνουμε μια εναλλακτικό ψηφίσμα ώστε να είναι πιο υπεύθυνη αυτή η πράσινη συμφωνία, πιο ρεαλιστική, πιο, με μεγαλύτερη συνοχή. Ειδικότερα αν λάβει κανεί υπόψη τι εκατοντάδε εκατομμύρια ευρώ που θα κινητοποιηθούν. Πολλοί σε αυτή τη συνέλευση εξακολουθούν να υποστηρίζουν μια ε, ελαφρόμυαλη ουσιαστικά συνένεση που θα ζημιώσει τους Ευρωπαίους και σε κοινωνικό και σε οικονομικό επίπεδο. Πρέπει να δείξουμε ευθύνη, ε, να σταθούμε στο ύψος της ε, ε, εκτίμησης που έχουμε προς τα οικολογικά θέματα. Ευχαριστώ, ζητώ συγγνώμη, δεν σας είδα κύριε Χάναν. Έχετε τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν 50 χρόνια λιοντάρια, τίγρης, λύκοι βρίσκονταν σε κίνδυνο. Σήμερα τα λιοντάρια παραμένουν υποπίεση. Οι τίγρες έχουν ε, σχεδόν εξαφανιστεί και οι λύκοι ε, ε, ζουν μια χαρά. Γιατί, Γιατί ζουν σε πλούσιες χώρες, ενώ τα άλλα ζουν σε φτωχές χώρες. Το καλύτερο πράγμα που μπορεί να συμβεί για το περιβάλλον είναι ο καπιταλισμός αγοράς. Ο Μάρξ το είπε ότι η φύση πρέπει να σε αντικείμενο εκμετάλλευσης. Ε, είδαμε τι έγινε στο Ανατολικό Μπλοκ με τις βιομηχανίες εκεί. Η θάλασσα της Αράλης έγινε μια έρημος, ένα σωρό μέρη ερημώθηκαν. Ε, παρότι έλεγαν στους ανθρώπους να μην πετάνε τι γόπε από τα πλοία. Η βιοπικιλότητα, η προστασία των ε, ειδών που κινδυνεύουν ε, είναι κάτι που, προστα... που δεν συνέβη σε χώρες που υπα... τα υπερασπιστήκαμε σε χώρες πλούσιες Εάν θέλετε να συντηρηθεί και η φύση, πηγαίνετε στους συντηρητικούς Ευχαριστούμε ο κύριος Βόντρα από το ECR. Ένα λεπτό, ευχαριστώ. Εκτός μικροφώνου ο μιλητής. Για να εξοικονομήσουμε για να εξοικονομήσουμε πόρου να διατηρήσουμε τα ύδατα ε, και να συντηρήσουμε τα δάση. Ε, πιστεύουμε ότι το κείμενο αυτό είναι υπερβολικό και δεν έχει καθόλου ρεαλιστικού στόχου. Γι' αυτό δεν μπόρεσα να το υπερψηφίσω ο στόχο μείωση ε, μέχρι το 2030 δεν είναι καθόλου ρεαλιστικός, ε, ενώ η πόρη που ε, δεσμεύτηκε να δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον προϋπολογισμό είναι γελίο ποσό, είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Οι τροπολογίες που υποβάλαμε για να στηρίξουμε την πυρηνική ενέργεια που θα μπορούσε να βοηθήσει την μετάβαση διότι θα, θα χρειαστούμε ε, πυρηνική ενέργεια για τη θέρμανση, για παράδειγμα. Ε, οι τροπολογίες αυτές καταψηφίστηκαν και γι' αυτό καταψήφισα και το ψήφισμα. Κυρίες και κύριοι, είμαι κάθετα εναντίον της μιας Πράσινης Συμφωνίας και όχι μόνο γιατί πρόκειται για ένα παράδοξο έγγραφο αυτού του νέου ρεύματος που υποστηρίζεται από ένα πνεύμα νεύρωσης υποκριτικής, φαρισαϊκό είναι. Μα πώς τολμάτε να δίνετε αγώνες προς αυτό το μέτωπο. Πριν από κάποιους μήνες ψηφίσαμε τα μέτρα για τις οδικές μεταφορές με τα άδεια φορτηγά που οδηγούν στην ανεργία τους βούλγαρους φορτηγατζίδες Τώρα λέτε ότι θα πρέπει να σταματήσει η εξόρυξη άνθρακα στην Ανατολική Ευρώπη. Όλα αυτά τα ψηφίζουμε, αλλά από την άλλη μεριά δεν υποστηρίζουμε την πιο οικολογική μορφή ενέργειας που είναι η πυρηνική ενέργεια. Η ολική ενέργεια, λέτε, και ταυτόχρονα βλέπουμε υποδομές, βλέπουμε όλα τελικά να γίνονται μία επεργολαβία προς την Κίνα. It's your Νίνα Τζιλ, είναι η σειρά σας, λέει η πρόεδρος. Εγώ είμαι αναφαντών υπέρ της νέας πράσινης συμφωνίας γιατί πρόκειται για μεγάλη πρόκληση, τόσο μεγάλη που χρειαζόμαστε μια μεγάλη επανάσταση και να μην περιστούμε σε αυτό που κάνουν οι κυβερνήσεις. Το σημαντικό είναι τι κάνουμε εμείς και τι σπρώχνουμε τον κόσμο να κάνει. Βέβαια το βάρος, την ύφη δεν θα πρέπει να την πληρώσουν οι πιο φτωχοί. Να εξασφαλίσουμε ότι οι λαϊκιστές δεν θα εκμεταλλευτούν, δεν θα χρησιμοποιήσουν τον φόβο της αλλαγής που έχει ο κόσμος γιατί έτσι εμείς θα πρέπει να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια για τη βιωσιμότητα στον πλανήτη στην ΕΚΟΝ δούλεψα σχετικά. Μπόρεσα να λάβω κάποιες πρωτοβουλίες όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά. Έχω και την έκθεσή μου για τα κριτήρια, τα benchmarks και αυτά και πάντως είμαι πολύ χαρούμενη και ψήφισα υπέρ. Σας ευχαριστούμε, λέει πρόεδρος. Ε, ευχαριστούμε. Και επεξηγήσεις ψήφου συνεχίζουμε τώρα ψήφισμα όσον αφορά την εφαρμογή και την παρακολούθηση των διατάξεων σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών στη Συμφωνία Αποχώρηση. Πρώτο ομιλητή είναι ο κ. Σκέλε. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Oh, I'm very sorry. I didn't realize that he left. Α, έφυγε. Δεν το κατάλαβα. Πήρε το λόγο και στην προηγούμενη συζήτηση. Τζάκι Jones τώρα, όπως και πριν, εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών.